εντός 24 ωρών και με βάση το άρθρο 105 οι συστάσεις λοιπόν θεωρούνται ότι ενεκρίθησαν και θα δημοσιευθούν μαζί με τα κείμενα που θα δημοσιευθούν αύριο 25 Δεκάτου 2017. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Έκθεση στάς. Χορήγηση απαλλαγής 2015 για το Γενικό Προϋπολογισμό. Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να δώσω το λόγο λοιπόν αρχικά